Επαναλαμβάνεται η περίοδο συνόδου που διακόψει 26 Νοεμβρίου. Τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26 Νοεμβρίου διατίθενται. Έχετε αντιρρήσεις, ενστάσεις,